Βάσει του άρθρου 3, παράγραφο 4 του ιστορικού κανονισμού, η Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων στη συνεδρίασή τη, που έλαβε χώρα στι 11 Ιουλίου του 2011 επαλήθευσε τα διαπιστευτήρια και επιβεβαίωσε ε, την εντολή των εξής βουλευτών Τάρια Κρόνμπερκ και Δημήτριος Δρούτσας ε, με ισχύ από την 22 Ιουνίου του 2011 και για τον κύριο Φρανκ Προύστ ε, με ισχύ από την 23 η Ιουνίου του 2011. Τρεις συνάδελφοι λοιπόν, σας, ε, ε, αυτοί οι τρεις ε, συνάδελφοι δικαιούνται συγχαρητήρια ολοκλήρωσαν τη διαδικασία και η Ολομέλεια καλείται να εγκρίνει την επιβεβαίωση των εντολών αυτών των τριών βουλευτών. Δεν βλέπω κάποια αντίρρηση. Είστε πλέον πλήρη μέλη. Ε, έχετε πλήρη δικαιώματα βουλευτέ βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Συγχαρητήρια. Βλέπω ότι από την ε, διάφορες ομάδες, την ΚΟΕ, τους Πρασίνους και τους φιλελευθέρους ε, έχουν κατατεθεί οι προτάσεις για διορισμούς για τις επιτροπές. Θα συνήψουμε τη